Herr Präsident! Die Sitzung ist äh, wieder aufgenommen. Αρχίζει και πάλι η συνεδρίαση. Παρακαλώ, καθίστε στις θέσεις σας. Περνούμε τώρα στον τρίτο γύρο της ψηφοφορίας. Νέες υποψηφιότητες για τον τρίτο γύρο για το αξίωμα του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν έχω λάβει δυνάμει του κανονισμού. Διατηρούνται οι υποψηφιότητες όπως είχαν και στο δεύτερο γύρο. Παρακαλώ τώρα τους κλητήρες να διανύμουν ψηφοδέλτια και φακέλους για την ψηφοφορία. Παρακαλώ τους ψηφοδέλτες να έρθουν στη θέση τους στις κάλπες. Οι ψηφοδέλτες παρακαλώ να λάβουν τις θέσεις τους.